Good morning everybody. Καλημέρα σας. Σας ε, χαιρετίζω και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα έχω τέσσερις ομιλητές και θα παρουσιάσουμε τα πορίσματα της ε, ε, αποστολής της Τρόικα στην Ελλάδα. Ε, είναι εδώ ο κύριος Σφόμποντα, επικεφαλής πολιτικής ομάδας, ο κύριος Κιόμπελς, πρώην Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, η Ελίζα Φερέρα από το Λουξεμβούργο και ο καθηγητής που ήταν και καθηγητής μαθηματικών και ο Ιβάλο Κάλφιν από την Βουλγαρία που είναι ε, πρώην ε, ε, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπεύθυνο εξωτερικών σχέσεων. Θα μιλήσει πρώτα ο Χάνες και μετά ο Ρομπέρο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της τριμερούς ομάδος στην Ελλάδα, θα μιλήσει στη συνέχεια. Ξέρετε <clears throat> ότι ζήτησα από τη Λίλιαν και τους δύο κυρίους να πάνε στην Ελλάδα και να <clears throat> καταρτήσουν μία τριμερή ομάδα για την ανάπτυξη και ε, το, την απασχόληση διότι η πραγματική τρόικα, η επίσημη τρόικα δεν ήταν ε, και τόσο επιδεκτική και ε, συζητήσιμη με τους πολίτες και επιπλέον δεν είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική αν δείτε όλες τις προβλέψεις της επισήμου Τρόικας την χάνουν, πρέπει να διορθωθούν και πολλές φορές μία-δύο εβδομάδες αφού δημοσιεύθηκαν αυτές οι προβλέψεις. Οπότε αυτή η πολιτική τρομερής λιτότητας και μειώσεως των εισοδημάτων των συντάξεων, των ημερομισθείων δεν είναι πολύ αποτελεσματική εκτός του ότι είναι αντιλαϊκή και αντικοινωνική ε, δεν φέρει και αποτελέσματα όπως θα πούν οι συνάδελφοι στη συνέχεια. Οπότε το πρώτο βασικό θέμα είναι να πούμε στην ε, ε, Τρόικα ότι πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ζήτησε από τον, από τον Πρόεδρο και την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Τρόικα ή στο Κοινοβούλιο για να εξεταστεί από το κοινό στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων διότι όπως σας είπα δεν είναι δυνατόν να πέφτει κανείς ε, σαν ε, ε, τα κοράκια πάνω σε μία χώρα και να την αφήνει φεύγοντας σε πλήρες χάος. Αυτή την πολιτική δεν την αποδεχόμαστε και πρέπει βεβαίως να βρούμε και εναλλακτικέ λύσεις και όπως θα σας πει ο κύριος Γκέμπελς και οι συνάδελφοι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί και στην Ελλάδα και αυτό είναι το δεύτερο θέμα η συζήτηση πρέπει να γίνει με τον ελληνικό λαό και τα ελληνικά θεσμικά όργανα όχι μόνο εκ των άνω αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχει συνεργασία. Οι Έλληνες ξέρουν για την οικονομία τους τι μπορεί ε, να είναι αποτελεσματικό, ποιες είναι οι δυνατότητες ε, και πώς πρέπει να γίνουν. Όντως πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, πρέπει αλλά οι σωστές μεταρρυθμίσεις, αυτές που θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα επισέλθω σε άλλε λεπτομέρειες διότι αυτά θα παρουσιαστούν από τους συναδέλφους αλλά ένα θέμα που πρέπει να σας πω και το συζήτησα και με τον πρέσβη σχετικά με την φοροδιαφυγή ε, και τις φορολογικές συμφωνίες είναι απαράδεκτο οι φτωχοί στην Ελλάδα να φορολογούνται με υψηλότερους ε, συντελεστές από ό,τι στο παρελθόν και να υπάρχει φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό προς την Ελβετία, υπάρχει συνεργασία η οποία ελπίζω να ολοκληρωθεί ο νουπο και υπάρχει ήδη μία συμφωνία μεταξύ των αρχών της Ελβετίας και της ε, Μεγάλης Βρετανίας που ε, έχει ε, πάρει το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα μπορέσει να γίνει μεταξύ των ελβετικών αρχών Αρχών και της Ελλάδος ασχέτως από τις ενδεχόμενες μελλοντικές ε, συζητήσεις περί Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις με την Ελλάδα θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσουμε διορθώσει η Τρόικα τον ε, προσανατολισμό της ε, και για ορισμένες προτάσεις θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται θα γίνει μια μελέτη η οποία έχει γίνει για το αποτέλεσμα της ε, Τρόικα και των συμβουλών που έχει δώσει στο παρελθόν θα να μορφώσουμε τη μελέτη αυτή που έχει καταρτιστεί από ένα γερμανικό Ινστιτούτο δεν είναι δηλαδή το τέλος της εργασίας μας για την Τρόικα αλλά η αρχή και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση να δούμε πώς θα αυξήσουμε τις πραγματικές επενδύσεις πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα διότι δεν είναι δυνατόν όλοι να ε, ε, τα ξέρουμε όλα μετά από λίγες εβδομάδες παρακολουθούν θύσεως της Ελλάδες έχουν γίνει λάθη στην Ελλάδα, μπορούν να διορθωθούν και θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι στο παρελθόν και δίνω τώρα το λόγο στον Ρομπέρ Γκέμπελς. Ευχαριστώ Χάνες. καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους στην ανεπίσημη αυτή αντιπροσωπεία τον Ήβαϊλο και την κυρία Φερέιρα που θα παρέμβουν και αυτοί αργότερα αν χρειαστεί. Εμείς δεν θελήσαμε να κάνουμε μια επίσημη αναφορά και έκθεση με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από την έκθεση της Επιτροπής. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά εξετάζοντάς τα βλέπουμε ότι πάντα τα ίδια ακούγονται, τα εύκολα. Πρέπει να σωθεί η Ελλάδα με εσωτερική υποτίμηση. Αλλά στο κείμενο της Κομισιόν και τα κείμενα του Δουνουτού βλέπετε ότι δεν επετέχθη ποτέ αυτός ο στόχος. Μάλιστα, μείωσαν τους μισθούς, μείωσαν τις συντάξεις, έκοψαν τις κοινωνικές παροχές, αλλά ταυτόχρονα μείωσαν και την αγοραστική δύναμη του λαού και για να εξισορροπηθεί ο προϋπολογισμός η Τρόικα πρότεινε την αύξηση των φόρων ιδίως του ΦΠΑ με αποτέλεσμα καθώς μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του κόσμου να μην μπορεί να δαπανίσει ό,τι ανέμενε να δαπανίσει και τα έσοδα της κυβέρνησης επομένως ιδιαίτερα από το ΦΠΑ έπεσαν παρά την αύξηση του ποσοστού. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Αν μειώσει κανείς τους μισθούς, τις συντάξεις και τα λοιπά, τότε διαθέτει λιγότερους πόρους για την κοινωνική ασφάλιση και τώρα υπάρχουν καινούργιες τρύπε και λύματα 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση που είναι άμεσο αποτέλεσμα της λεγόμενης αυτής εσωτερικής υποτίμησης. Μόνο μείωση των μισθών. Τίποτα δεν έγινε για να σταματήσει η αύξηση των τιμών. Δεν πάγωσαν οι τιμές, τίποτε τέτοιο. Ο πληθωρισμός μάλιστα αυξάνεται και ξεπερνάει τον μέσο όρο της Ένωσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα η Τρόικα δεν πέτυχε αυτά που σκόπευε να πετύχει και αυτά που επέβαλε στη Ελληνική Βουλή πολιτικούς και λαό. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο Πρέπει η Τρόικα να είναι υπόλογη και υπεύθυνη και γι' αυτό ζητούμε να έρθει, να έρχεται τακτικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πρώτη τέτοια συνάντηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την Τρίτη σε κοινή συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης και της Οικονομικής και Νομισματικής. Επίσης λέμε ότι χρειάζεται, πρέπει, να δούμε και κοινωνικά τι έγινε. Ζητούμε λοιπόν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής πλατφόρμας, διότι υπάρχει διάλογος μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων στην Ελλάδα, οι οποίοι συμφώνησαν, τα δύο αυτά μέρη συμφώνησαν, να γίνει τριετές πάγωμα των μισθών τριετές πάγωμα των μισθών. Η Τρόικα όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό και ζήτησε μείωση περαιτέρω των μισθών κατά 22%. Επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικά μέτρα για την οικονομία γιατί το Δουνουτού και τα έγγραφα της Τρόικας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δείχνουν ότι κάθε δύο-τρεις μήνες γίνεται προσαρμογή, αναπροσαρμογή για πολύ, έναν πολύ απλό λόγο γιατί θεωρούν ότι αυτή η εσωτερική υποτίμηση των μισθών θα έφερνε περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Δεν έφερε όμως τίποτα τέτοιο μόνο μείωση της ζήτησης, της εσωτερικής ζήτησης στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Τα τελευταία πέντε χρόνια ή μάλλον στο τέλος αυτού του έτους η Ελλάδα θα είναι πάλι σε ύφεση και σύμφωνα με επίσημους αριθμούς της Τρόικας και του Δουνουτού μέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα θα έχει ύφεση της τάξης του 22,6% τουλάχιστον. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι μηχανιστικά θα αυξηθεί η σχέση χρέους με ΑΕΠ. Η ύφεση αυτή πρέπει να καταπολεμηθεί επιγόντως η Ελλάδα δεν θα σωθεί παρά μόνον εάν επανέλθει στην ανάπτυξη και άρα και στην απασχόληση. Το πρώτο κατεπήγον μέτρο είναι πλήρης ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πληγεί πάρα πολύ πρώτον είχαν πολλά ελληνικά, ομόλογα του ελληνικού χρέους και το κούρεμα που έγινε τελευταία τους δημιούργησε πολλές απώλειες. Έπειτα πολλά χρήματα έφυγαν από τη χώρα, 70 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται και η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών είναι καταστροφική. Αυτό φαίνεται σε όλα τα έγγραφα της Κομισιόν του Δουνουτού εδώ και μήνες. Και ο ηγέτης της Ομάδας Εργασίας για την Ελλάδα πριν από έξι μήνες ζήτησε, είπε ότι το πιο επίγον μέτρο θα ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τώρα λένε ίσως το Σεπτέμβριο να γίνει κάτι. Αν όμως οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν πολύ γρήγορα, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στις αγορές. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία υπηρεσία για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που να είναι ο άμεσος συνομιλητής των ιδιωτών ή δημοσίων αρχών που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να, να διευθύνεται από κάποιον Έλληνα με τη βοήθεια εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Δουνουτού και της κυβέρνησης, καθώς και των κοινωνικών εταίρων. Η ιδέα αυτή εμφαίνεται και σε ένα εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν που κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχω αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να το παραπέμψω σε αυτό προτείνεται εκεί αμέσως βραχυπρόθεσμα να δημιουργηθεί ένα εργαλείο ρευστότητας 300 με 500 εκατομμύρια για να υπάρξει εγγύηση των δανείων των τραπεζών. Ακόμα και η Κομισιόν λοιπόν αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μια τέτοια επενδυτική υπηρεσία χωρίς να εξετάζουμε τι λέει η Standard και Poor's και η Moody's και τα λοιπά. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει αμέσως να αρχίσει η εφαρμογή των 181 προγραμμάτων ή σχεδίων που έχουν ταυτιστεί από την ομάδα εργασίας της Κομισιόν υπό τον κύριο Ράιχενμπαχ που γενικά δουλεύει καλά και ταύτισε 180 σχέδια που πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως με χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων και μερικά χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Πρώτο θέμα λοιπόν η αναδιάρθρωση των τραπεζών. Γενικότερα εμείς οι σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αυξήσει την κεφαλαϊκή της βάση κατά τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια για να μπορεί να χρηματοδοτήσει περισσότερες επενδύσεις και στην Ελλάδα και αλλού στην Ευρώπη. χρειάζονται επενδύσεις παντού. 10 δισεκατομμύρια για 27 κράτη-μέλη δεν είναι τίποτα βέβαια. Αλλά αυτό θα μπορούσε να δώσει στην ΕΤΕ και στην ευρωπαϊκή οικονομία κάποια ανάσα τουλάχιστον προσωρινή. Έπειτα όπως είπε και ο Χάνες πριν υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Όλοι ξέρουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μακρά παράδοση φοροδιαφυγής. Οι εφοπλιστές έχουν το μεγαλύτερο στόλο του κόσμου αλλά πληρώνουν σχεδόν μηδενικούς φόρους στην Ελλάδα επειδή η έδρα τους, τα γραφεία τους είναι επισήμως σε κάποια μυστήρια νησιά. Η ελληνική κυβέρνηση προς το παρόν συζητάει με την Ελβετική για να υπάρξει κάποια συμφωνία όπως, μεταξύ, όπως με τη Γερμανία και την ε, Βρετανία. Αυτό είναι επίσης απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η συμφωνία πρέπει να υπάρξει, να υπογραφτεί και να εγκριθεί, να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο φέτος ώστε να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Και μετά επίσης χρειαζόμαστε απολύτως στην Ένωση προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και υποστήριξης της ανάπτυξης. Ήδη στην ομάδα μας κάναμε, διατυπώσαμε λεπτομερείς προτάσεις και εναλλακτικέ λύσεις μέσω συντονισμένων ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων με εργαλεία όπως τα ευρωομόλογα και φυσικά τον φόρο των δοσοληψιών ως καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτές είναι ορισμένες ιδέες που πιστεύουμε ότι είναι ζώτικες για να επανέλθει η Ελλάδα σε έναν αναπτυξιακό δρόμο και να βγει από την ύφεση. Αυτό είναι απόλυτη αναγκαιότητα, αλλιώς οποιαδήποτε βοήθεια προσφέρεται θα αποβεί μάταιη. Ευχαριστούμε, αναμένουμε ερωτήσεις. Ωραία, βλέπω εδώ. Παρακαλώ να λέτε και ποιοι είστε και για ποιο όργανο εργάζεστε. Ο Ντέτλερ Φέχνερ από την Πόρσεν Zeitung αναφερθήκατε ε, για το ERB και να αυξηθεί ε, η κεφαλαϊκή βάση. Είστε σε επαφή με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη και έχετε την εντύπωση ότι αυτοί θα συνενέσουν Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο νέος πρόεδρος του ERB, ο κύριος Βέρνερ Χόιερ, ε, προτείνει να αυξήσει την κεφαλαϊκή του βάση. Οπότε δεν νομίζω δεν νομίζω ότι οι λίγες κυβερνήσεις που διοικούνται από σοσιαλιστές στην Ευρώπη αποτελούν εμπόδιο. Αυτό που πρέπει να ε, αυτούς που πρέπει να πείσουμε είναι τα μεγάλα κεφάλια, η Γερμανία, η Γαλλία, ενδεχομένως και την ε, Μεγάλη Βρετανία η οποία δεν μπορεί συνέχεια να αποφεύγει τις ευθύνες της για την Ευρώπη και όταν μιλάμε για τα ευρωομόλογα, ήδη υπάρχουν ευρωομόλογα. Αυτά είναι τα ομόλογα τα οποία εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως, η οποία εγγυούνται οι 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πέρυσι η τράπεζα αυτή εξέδωσε νέα δάνεια για 70 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν είναι μικρό ποσό και εφόσον εγγυώνται από 27 κράτη-μέλη και έχουν ε, βαθμολογηθεί με τριπλό αλφα χρειάστηκε να πληρώσουν μεταξύ 3-2 γύρω στο 2,5% επιτόκιο στη διεθνή αγορά πράγμα το οποίο δεν είναι κακό είναι κοντά στα Bundesbriefe της ε, γερμανικής κυβερνήσεως. Άλλη ερώτηση. Με ενδιαφέρει πολύ η ιδέα ότι η Τρόικα πρέπει να είναι υπόλογη και υπεύθυνη. Να λογοδοτεί δηλαδή. Αν κατανοώ καλά θα έρθει η Τρόικα στο Κοινοβούλιο ενώπιον δύο επιτροπών σε κοινή συνάντηση. Κοινή συνάντηση. Ερωτώ λοιπόν σε τι βασίζεται αυτό. Κανονικά η Κομισιόν αναφέρει, είναι, συζητάει με το Κοινοβούλιο. Δημιουργείται έτσι κάποιο καινούργιο είδος πρωτοκόλλου, μια καινούργια διαδικασία. Πώς θα λογοδοτεί ακριβώς. Θα έρθουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις, αλλά αυτό σημαίνει ότι λογοδοτούν και όλα. Εδώ υπάρχει το αίσθημα ότι ξεπερνούν κατά πολύ τις δικαιοδοσίες τους με τις περικοπές μισθών συντάξεων και κανείς δεν ξέρει με τι ακριβώς βάση. Ναι, με την τελευταία σας φράση αναφέρεται ακριβώς το πρόβλημα. Και εμείς αυτό ρωτάμε. Ποιος έδωσε την εντολή στην Τρόικα να επιβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση τη μείωση των ελαχίστων μισθών και των συντάξεων. Ποιος. Το έθεσα το ερώτημα εξ ονόματος της ομάδας μου στην Ολομέλεια πριν από δύο μήνες και η απάντηση της Κομισιόν ήταν ότι η Ευρωζώνη, το Eurogroup το ζήτησε. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό, αλλά αυτό απάντησαν. Χρειάζεται λοιπόν εδώ κάποια σαφήνεια. Ποιος μιλάει εξ ονόματος της Ένωσης στη συνεδριάση της Τρόικας. Μπορούμε να ρωτήσουμε τους επιτρόπους, τον πρόεδρο του Eurogroup ή τον πρόεδρο του Εκοφήν οποιονδήποτε άλλον, αλλά νομίζω ότι οι λαμπροί αυτοί ανώτατοι υπάλληλοι που προσέρχονται στην, που πηγαίνουν στην Ελλάδα για μια εβδομάδα τα ξέρουν όλα και επιβάλλουν τέτοια ριζοσπαστικά μέτρα πρέπει και αυτοί να θεωρούνται υπόλογοι. Γι' αυτόν τον λόγο την επόμενη εβδομάδα θα τους φέρουμε σε αυτήν την κοινή συνάντηση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής Απασχόλησης και θα δούμε εκεί. Όπως βλέπετε και στο σημείωμά μας θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πίεση επί της Κομισιόν αλλά και των ανωτάτων υπαλλήλων που μιλούν εξ ονόματος της Ευρώπης. Εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε εκλεγεί από τους πολίτες. Όλοι αυτοί όμως έχουν διοριστεί απλώς. Ακόμη και αν είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι να εξυπηρετούν τους επιτρόπους, παρόλα αυτά πρέπει να είναι και αυτοί υπόλογοι. Αυτό προσπαθούμε. Ε, θα προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή, Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπόλογοι προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι έρχονται να εξηγήσουν τις πολιτικές τους. Ενώ στην περίπτωση της Τρόικα υπήρξαν πολλές μυστικές δραστηριότητες και καμιά ανάληψη ευθύνης. Οπότε όταν τους κάνουμε ερωτήσεις, άλλοι μας αποφεύγουν και μας λένε λόγω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θα ήμασταν τόσο αυστηροί αν ήταν μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα ήμασταν τόσο αυστηροί οπότε θέλω να δω αν υπάρχει μία ενοποιημένη θέση ποιος ευθύνεται για την αποτυχία των δραστηριών της Τρόικα διότι υπάρχει πάντοτε η πρόβληψη ότι όλα θα πάνε καλύτερα ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά και όλα αυτά έπρεπε συνέχεια να διορθώνονται ε, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για το μέλλον. Όχι μόνο αυτή η τρόικα αλλά και η δραστηριότητα και σε άλλες χώρες και στην Πορτογαλία και αλλού πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην αφήνουμε ε, ελεύθερου αυτούς ε, του κυρίους οι οποίοι κυκλοφορούν ε, και εγώ είμαι οικονομολόγος αλλά δεν θα τολμούσα να πάω σε μια χώρα και να του πω περικόψτε, περικόψτε, περικόψτε. Χρειάζεται κανείς να ξέρει τα συμφραζόμενα φαινόμενα. Ε, εάν γνώριζαν καλύτερα την Ευρώπη ίσως δεν θα συμπεριφέρονταν έτσι. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω αλλά θέσατε το θέμα των στρατιωτικών δαπανών στην Ελλάδα το ρόλο που παίζει δηλαδή στον προϋπολογισμό της φαίνεται ότι δεν έχει περικοπεί καθόλου ο στρατιωτικός προϋπολογισμός και ακούμε διάφορα τρομερά για αγορές υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων που τους τελευταίους μήνες ακούγονται και για δοσοληψίες Ελλάδας, Γερμανίας, για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Γιατί δεν περικόπτουν αυτές τις δαπάνες αντί για τα συντάξεις. Δεύτερο ερώτημα. Μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Τρόικας φαίνεται να είναι η κυριότερη προτεραιότητά της ότι όλα τα χρήματα καταρχήν θα αποπληρώνουν το χρέος και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αυτό το αμφισβητείτε, τους λέτε ότι δεν μπορείτε να λέτε σε μια χώρα ότι το επιτόκιο για εξυπηρέτηση του χρέους είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ευχαριστώ οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν περικοπεί και αυτό είναι πολύ καλό αλλά το περίεργο είναι ότι μερικές από τις χώρες μέλη που επέκριναν τόσο πολύ την ελληνική πολιτική πουλάνε όπλα στην Ελλάδα, η Γαλλία και η Γερμανία ας πούμε και συνεχίζουν να το πράττουν σε εποχή που είναι φανερό ότι τέτοιες πωλήσει αυξάνουν το πρόβλημα. Η, περικοπή των στρατιωτικών δαπανών είναι καλή γενικώ, αλλά δεν μπορεί μερικές χώρες από τη μια να επικρίνουν και από την άλλη να πουλάνε όπλα. Τώρα πρέπει να φύγω δυστυχώς, θα απαντήσουν οι υπόλοιποι. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της βοηθείας το οποίο δόθη από την Ευρώπη και την Ευρωζώνη προς την Ελλάδα ήταν μια βοήθεια που απέβλεπε να βοηθωθούν οι χώρες δωρητές όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν όταν είχαν βοηθήσει να αποφύγουν οι τράπεζες τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες να ζημιωθούν από την ελληνική χρεοκοπία οπότε γι' αυτό η ομάδα των ε, σοσιαλιστών δημοκρατών ε, ηγείται αυτής της προσπαθίας ε, ίσως δεν βλέπετε αρκετά μέσα στο σημείωμα που ετοιμάσαμε τι εργασία γίνεται αλλά θέλω να έχω σαν ε, ε, σαν μάρτυρα τον πρόεδρο του ε, Eurogroup τον Ζων Κλοβιούντ Γιούνκερ που είναι φίλος μου αλλά και ανταγωνιστής μου είμαστε από την ίδια χώρα όπως ίσως ξέρετε και σε μία συνέντευξη στην ελληνική εφημερίδα Καθημερινή είπε και λέω ότι αν θέλετε η χώρα να ε, επανέλθει ε, στη σωστή πορεία θα πρέπει να υπάρχει ε, μία φορολογική βελτίωση αλλά και κίνητρα αναπτυξιακά. Στην Ελλάδα εμείς δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί στο θέμα της ανάπτυξης και υπερβολικά δυνατοί σε φορολογικά και αυτό ακριβώς συνέβη. Δηλαδή η Ευρώπη και το Δούνου του επέμειναν πάρα πολύ για τη φορολογική βελτίωση με ε, εσωτερική υποτίμηση, με μείωση των μισθών χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ε, δώσουν νέα κίνητρα στην ελληνική οικονομία. Και η χώρα αυτή εδώ και πέντε χρόνια πάει από τη μία ύφεση στην άλλη έχει όντως σοβαρά προβλήματα και αυτό λέμε και εδώ στο εγγραφό μας ότι πρέπει να επιμείνουμε στις επενδύσεις να εισρεύσει ζωντανό χρήμα κατά τρόπον ώστε η οικονομία να λειτουργήσει η ανεργία να μειωθεί να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ε, υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα ε, υπάρχει και περισσότερο αντικείμενο προς φορολόγηση, ε, πληρωμή ε, κοινωνικών εισφορών κτλ. Χωρίς ε, ανάπτυξη τίποτα δεν θα μπορέσει να γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει καμιά τελευταία ερώτηση. Πολύ σύντομα η Σάρα Κόλινς από το Europolitis, μία διευκρίνηση. Ε, ξέρετε ε, πόσα χρήματα σε στρογγυλά θέλετε να αντλήσετε προς την Ελλάδα και επειδή είναι και η Ελίζα Φερέρα και η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την σοβαρή ε, ύφεση οπότε προτείνεται την ίδια λύση για την Πορτογαλία και για την Ιρλανδία μέσω επενδύσεων. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι όλης της Ευρωζώνης και της δυνατότητάς της να επιβιώσει το, τις κρίσεις. Αφού αν συστήσουμε σε κάθε χώρα που έχει πρόβλημα να λάβει μέτρα που καταλήγουν σε ύφεση, τότε δεν θα έχει κανένα πλεόνασμα και δημιουργούμε έναν κύκλο ύφεση που αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο και τις χώρες αυτές και ολόκληρη την Ευρωζώνη και τελικά την Ευρώπη ολόκληρη. Είναι λοιπόν σοβαρό το πρόβλημα και νομίζω ότι αυτά που ζητάμε τώρα για την Ελλάδα τελικά στοχεύουν στην έξοδο από αυτόν τον φαύλο κύκλο για να υπάρξει ανάκαμψη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι δυνατόν αν υπάρξει βέβαια η απαραίτητη πολιτική θέληση και συμφωνία επί των πολιτικών στόχων αλλαγής μιας πολιτικής που δεν έχει πετύχει πριν φτάσουμε στην τελική και αναπόφευκτη καταστροφή για να επανέλθω στο πρώτο τμήμα της ερώτησης σας δεν έχουμε κανένα σχέδιο ολοκληρωμένο λέμε απλώς να σταθεροποιηθούν οι τράπεζες για να μπορέσουν να ξαναλάβουν την κανονική τους λειτουργία της χρηματοδότησης της οικονομίας. Τα 181 προγράμματα που έχουν ταυτιστεί από την ειδική η ομάδα εργασίας της Κομισιόν και για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια από τα διορθωτικά ταμεία έχουν προβλεφθεί για την Ελλάδα. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δεν απορροφώνται. Αν χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά που ήδη έχουν εγκριθεί, θα ήταν ήδη σημαντικό. Και επίτα ζητάμε η ΕΤΕ να είναι λίγο πιο δραστήρια για να χρηματοδοτήσει περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί πάρα πολύ από τη συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας εδώ και πέντε χρόνια 200.000 θέσεις εργασίας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Πριν ήδη ξεσπάσει η έκδηλη κρίση. Πάντα χρειάζονται βέβαια χρήματα και δεν μπορούν πάντοτε όλα αυτά τα χρήματα να είναι δημόσιο χρήμα από την Ένωση. Υπάρχει θέση και για ιδιωτική χρηματοδότηση και τμήμα των 75 δισεκατομμυρίων που έχει φύγει από την Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει και να επανεπενδυθεί στην ελληνική οικονομία εφόσον μάλιστα αρχίζουν και άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Ξαναλέω όμως ότι το κλειδί για όλα αυτά όπως θα έλεγε και ο Μπιλ Κλίντον είναι απλώς η οικονομία δηλαδή δεν μπορούμε να τα καταστρέφουμε όλα και μετά να λέμε «Α, υπάρχει ύφεση». Ωραία. Και με αυτό τελειώνουμε. Αν υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τότε διμερός ιδιωτικός να τα θέσουμε. Υπάρχει εδώ και το έγγραφό μας. Σας ευχαριστώ όλους για την προσέλευσή σας.